Colleagues, ladies Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία αρχίζουμε. Οφείλεται στο ότι όταν καταφθάσαμε ακόμη συνεχιζόταν η προηγούμενη συνεδρία και δεν είχαμε την αίθουσα στη διάθεσή μας, γι' αυτό ε, αργοπορήσαμε. Βέβαια δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για ποιο λόγο μια προβλεπόμενη συνεδρίαση επιτροπής δεν ε, μπορεί να διεξαχθεί ε, διότι δεν είναι έτοιμη εγκαίρως ε, η αίθουσα. Αλλά ήθελα να σε εξηγήσω την κατάσταση. Ας αρχίσουμε με την έγκριση του σχεδίου ημερησία διατάξεως, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ε, εγκρίνεται με τις ακόλουθες ε, αλλαγές. Σημείο 11. Εξέταση ερώτηση για προφορική απάντηση προ το Συμβούλιο για τι Εμπορικέ Σχέσει ΕΕ Καναδά. Ακυρώνεται, διαγράφεται αυτό το σημείο. Σημείο 18 το σχέδιο έκθεσης του κ. τα μεταβατικέ ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μέλων και τρίτων χωρών αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 12 και 13 Απριλίου δηλαδή κατόπιν αιτήματος του εισηγητή και σημείο 31 για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση αυτό το σημείο θα το εξετάσουμε το πρωινό της 16 6η Μαρτίου, δηλαδή αύριο το πρωί. Το σημείο τώρα 25, ε, κατόπιν ετοίματος του. Ε, συγγνώμη, θα εξεταστεί αύριο το πρωί κατόπιν ετήματο του συγητή του κυρίου Γιάννη Ξαντό. Πριν προβώ στι ανακοινώσει ε, του Προέδρου, θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για την τραγουδία που ζει η Ιαπωνία. Η απώλεια ανθρωπίνων ζώων και οι καταστροφικές ε, υλικές ε, ζημιές ε, νομίζω απαιτούν ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ. Thank Ανακοινώσεις. Είναι στο διαδίκτυο το περιεχόμενο της συνεδριάσεώς μας, εκτός βέβαια του τμήματος κυκλισμένων των θυρών, όπου γίνεται η συνεδρία των συντονιστών. Ο κύριος Κάσπαρη, κύριε Πρόεδρε. Για το σημείο 1 έγκριση της τη διάταξης, αν μπορώ να επανέλθω, μετά τα καταστροφικά γεγονότα της ε, Ιαπωνίας, είναι πολύ δύσκολο να συζητήσουμε τα σημεία 9 και 10. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι να αφαιρέσουμε τα σημεία αυτά την ημέρησια διάταξη και ενδεχομένως αν η κατάσταση που κινδυνεύει να επιδεινωθεί θα έπρεπε να συζητηθεί στην ε, Ολομέλεια με ψηφίσματα, όχι εξ ονόματο τη Επιτροπή μα, αλλά καλύτερα εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό προτείνω τα σημεία 9 και 10 να αφαιρεθούν από την ημέρηση διάταξη. Ναι. Συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες για αυτή τη διαδικασία. Ο Μάρτιν. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε πάντα επίγνωση των συνδικών κάτω από τις οποίες λαμβάνουμε το λόγο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Από ό,τι καταλαβαίνω ο Ντάνιελ Κάσπαρη δεν θέλει να αναβάλει το θέμα αυτό, απλώς να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων στην Ολομέλη για τη διατύπωση, ε, χωρίς να συζητήσουμε σήμερα, κάτι το οποίο νομίζω ότι το να μην συζητήσουμε σήμερα είναι απόλυτα λογικό και εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ε, συμβαστική λύση να μην το θέμα στην ημέρησια διάταξη ώστε να δώσουμε κάποια συμβολή στη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας χωρίς φυσικά να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Τα σημεία λοιπόν 9 και 10 δεν θα βρίσκονται στη σημερινή μας ημερησία διάταξη. και ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες θα μπορέσουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να συγκλίνουν σε κάποιο κοινό κάποια κοινή διατύπωση και την προφορική ερώτηση με το ψήφισμα. Ανακοινώσεις τώρα. Έχουμε κάποια, κάποια αλληλογραφία και τα μέλη που ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε στοιχείο της αλληλογραφίας μπορούν να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την ε, γραμματεία. Δεν έχουμε βουλγαρική διερμηνία, λέει ο πρόεδρος, αντίθετα από την πραγματικότητα, αλλά θα είναι διαθέσιμη αύριο. Μάλλον αύριο δεν θα έχουμε βουλγαρική διερμηνία, γιατί σήμερα υπάρχει βουλγαρική διερμηνία, αλλά αύριο δεν θα υπάρχει. Συγγνώμη που δεν διάβασα σωστά τις σημειώσεις μου. Σε σχέση τώρα με το θέμα της ε, χρηματοδοτικής βοήθειας προς τη γεωργία, μετά την εφαρμογή των νέων εφαρμοστικών κανονισμών, θα χρειαστούν κάποιες τεχνικές προσαρμογές σε αυτή την πρόταση που ενεκρίθη από την Επιτροπή μας τον προηγούμενο μήνα με απλοποιημένη διαδικασία χωρίς ε, τροπολογίες. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νέα συμβουλευτική διαδικασία τη στιγμή που έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αυτός κανονισμός. Προβλεπόταν να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου, αλλά έχει αναβληθεί η ψηφοφορία γιατί η Κορεπέρ δεν μπορεί μέχρι τις 16 Μαρτίου να επικυρώσει το ότι συμφωνούν με τις τεχνικές αυτές προσαρμογές και οι 16 είναι οι προθεσμίες της τροπολογίας. Αν το Συμβούλιο λοιπόν θέλει τη νέα διαδικασία εξέτασης και όχι τη διαδικασία συμβουλευτικού χαρακτήρα, ο Πρόεδρός μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο εξ της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ζητώ λοιπόν να έχω αυτή την εξουσιοδότηση από εμάς με Υ. Έχετε κάποια αντίρρηση. Ελπίζω τώρα το Συμβούλιο δεν θα ζητήσει κάτι τέτοιο, αλλά αν το ζητήσει θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων την 1η Μαρτίου αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα παρακολούθησης με συμβουλευτικό χαρακτήρα για να παρακολουθήσει την πολιτική κρίση της ε, την σε Αιγύπτου και Λιβύης και να παρακολουθεί την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνολη περιοχή στο φως της αναθεώρησης της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής ε, για την περιοχή αυτή. Και η γραμματεία μας περιέχει και ένα αρμόδιο ο οποίος θα παρακολουθεί την διαδικασία της ομάδας αυτής παρακολούθησης. Τα μέλη της Επιτροπής μας που ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή αυτή προσκαλούνται να γίνουν μέλη ad hoc στην ομάδα παρακολούθησης. Παρακαλώ λοιπόν καταγράψτε και σημειώστε αυτό το σημείο. Ας πάμε στο σημείο ο David Μάρτιν δεν έχει να κάνει με αυτά που είπατε, αλλά αν μπορώ να το θίξω σε αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την αδυναμία των μελών της Επιτροπής μας να κάνουμε σωστά την δουλειά μας. Αύριο το απόγευμα έχουμε μια συνεδρία κυκλισμένων των θυρών με το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και θα μας μιλήσει για τις συμφωνίες τη Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου. Αλλά παρά το γεγονός ότι εσείς και η γραμματεία μας έχουν τα αντίστοιχα έγγραφα για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, τα μέλη της Επιτροπής μας δεν έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Αυτό κάνει απόλυτα δύνατο να έρθουμε σε μια συνεδρίαση αύριο το απόγευμα και να θέσουμε οποιαδήποτε ερώτηση που δεν είναι γενικού χαρακτήρα και θα λάβει γενικές απαντήσεις. Αν, δε... Αν θέλουμε να λάβουμε στα σοβαρά ε, αρμοδιότητες μας από τη Συνδίκη τη Λισαβόνα, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένε ερωτήσει και χωρίς τι απαραίτητε πληροφορίε, δεν μπορούμε να το κάνουμε και εγώ βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ματαιωτικό να είμαι μέλο αυτή τη επιτροπή. Well, since, Εφόσον μιλάτε για διαβαθμισμένα έγγραφα, ε, οι εφαρμοστέ κανόνες το προβλέπουν αυτό. Δηλαδή, ε, μόνο οι εισηγητέ και οι σκιώδει εισηγητέ έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, όχι τα υπόλοιπα ε, μέλη τη Επιτροπή. Αυτό προβλέπεται ε, στο καταστατικό. Αν θέλουμε τώρα τροποποίηση των κανόνων και πιστεύω ότι ίσω κάποιοι το επιθυμούν, πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να διαπραγματευτούμε τους νέους κανόνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί επί τούτο ad hoc σήμερα δηλαδή να αποφασίσουμε οτιδήποτε. Ε, απευθύνω έκκληση λοιπόν στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων αν το επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία τους ώστε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για τροποποίηση του κανονισμού που διέπει την πρόσβαση στα ε, διαβαθμισμένα έγγραφα, σε τέτοιου είδους έγγραφα. Σχόλια από τις πολιτικές ομάδες. Ο Ντέιβιντ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ε, αυτά προβλέπονται στους κανόνες. Ε, δεν ε, απευθυνόμουν ούτε σε εσά ούτε στη γραμματεία. Δεν το καταλόγησα σε εσά. Μιλούσα για τις συγκυρίες. Δηλαδή οι συντονιστές ναι, να συζητήσουμε ποιο τρόπο μπορούμε να τροποποιήσουμε τους κανόνες. Και πρόσφατα συζητούσαμε ένα μέλος του Κογκρέσου, τον είπα, που μου είπε ότι η διαπραγματευτική εντολή της Αμερικανικής Διοίκησης είναι προσβάσιμη σε όλα τα μέλη του Κογκρέσου, σε όλους τους γερουσιαστές, όχι μόνο αυτούς που έχουν επιληθεί της υπόθεσης εμεί όμως που είμαστε ενεργά μέλη της Επιτροπής ε, δεν έχουμε καν το δικαίωμα να τα δούμε τα έγγραφα, όχι μόνο να τα εξετάσουμε. Όχι να τα εξετάσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Πρόεδρος, είναι μια ευκαιρία για να ε, το μελετήσουμε το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά προϋπήρχαν οι κανόνες πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας Χρειάζεται λοιπόν νέο θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται τροποποίηση των ε, κανόνων. Αυτό πρέπει όμως να κάνει το Κοινοβουλίο, να παραβιάζει τους κανόνες, να τους τροποποιεί όταν αυτό επιθυμεί. Παρακαλώ, Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να στηρίξω αυτά που είπε ο Ντέβιτ Μάρτιν Ούτως ώστε να έχουμε πρόσφορη αποτελεσματική συζήτηση τα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το τονίζω, ε, δεν ξέρω αν πρέπει και κάποιος άλλος θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά τουλάχιστον οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, μα είναι λυπηρό, είναι απογοητευτικό να περιμένουμε την παρέμβαση του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης για να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Ε, δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση του Ντέβιτ Μάρτιν, πρόεδρος δεν ε, βρίσκω ότι έχει νόημα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα. Μπορείτε να το εγείρετε στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών, ούτω ώστε να καρποφορήσει η συζήτηση. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τους κανόνε, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχει βούληση, α το προσπαθήσουμε, αλλά μην ε, δηλώνετε έκπληκτη. Και εγώ θα πρότεινα να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών αλλά ήδη έχουμε συζητήσει τη συνεδρία των συντονιστών για το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα. Για μένα το βασικό είναι η δική μου πεποίθηση και θέλω να υποστηρίξω τον David Μάρτιν προς την κατεύθυνση αυτή, ότι δηλαδή κάθε μέλος της Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά τουλάχιστον της δικής μας Επιτροπής που είναι η αρμόδια για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ έχω πληροφορηθεί για την κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν υπάρχει, λένε ορισμένοι, κάποιος κανόνας στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Όχι, υπάρχουν σαφείς κανόνες κάτω από τους οποίους κάτω από συνθήκες εμπιστευτικότητος μπορούν να έχουν πρόσβαση βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου. Έχει προκύψει πολλές φορές από έγγραφα τα οποία δεν είναι δημόσια, τα οποία μας έχουν στείλει η Κομισιόν αυτά τα έγγραφα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Γι' αυτό θέλω να πω στους συναδέλφους ότι ναι μεν υποστηρίζω να, υπάρχουν, να υπάρχει πρόσβασή μας στα έγγραφα αυτά, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να επιληφθεί και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για το τι γίνεται στην περίπτωση που οι βουλευτές παραβιάζουν την εμπιστευτικότητα αυτών των ε, ε, εγγράφων και ποιες θα πρέπει να είναι οι ενδεχόμενες κυρώσεις για αυτή την περίπτωση Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώ θα κάνουμε εάν ορισμένοι συνάδελφοι παραβιάσουν αυτή την έννοια τη εμπιστευτικότητα η οποία πρέπει να ισχύει για τα έγγραφα αυτά. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Σούλτ, και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Υποστηρίζω αυτά τα οποία λέει ο κύριο Κασπάρη, γιατί είναι απόλυτα δικαιολογημένο αυτό το οποίο λέει ο κύριο ε, Μάρτιν θα πρέπει να επανέλθουμε στη συνεδρία των συντονιστών στο θέμα αυτό, αλλά καταρχήν εγώ υποστηρίζω απόλυτα την άποψη του David Μάρτιν. Right. Just let me that... Ωραία. Να προσθέσω ότι δεν μπορούμε μερός να τροποποιήσουμε τους κανόνες και η θέση μας έχει κάπως αποδυναμωθεί από μία σειρά διαρών που ε, επισυνέβησαν. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 3. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης των συντονιστών έχουν διανεμηθεί και θα θεωρηθούμε ότι εγκρίνονται αν δεν υπάρξουν ενστάσεις Σημείο 4. Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ. Η ΑΦΕΤ είναι επί τη ουσία αρμόδια επιτροπή. Εμεί ε, έχουμε συντάξει γνωμοδότηση, τη οποία συντάξει είναι ο συνάδελφο Εμίλιο τη ε, Ντεβάλε. Και σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο της γνωμοδοτήσεως Έχετε στο φάκελό σας το έγγραφο. Η Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία συμπεριλαμβάνει και ένα σημαντικό κεφάλαιο αφιερωμένο στο εμπόριο και σε επενδύσει. και συμπληρώνεται φυσικά και από τον έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διευθέτηση διαφορών. Πρόκειται λοιπόν για μια εμπορική συμφωνία με εγκάρσεις πολιτικές επιπτώσεις. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την απογοήτευσή μου που η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφάσισε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 110, κάτι που αποκλεί αδίποτε συνεργασία σε αυτό την έκθεση. Δηλαδή η Επιτροπή μας, που είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, δεν έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί επί τη Συμφωνία Τερικής Σχέσης και Συνεργασίας, ενώ ο εισηγητής μας ε, Μενέντες έχει τη δυνατότητα να προσαρτήσει αυτήν την συνοπτική αιτιολόγηση. σε διάφορες μικτές ε, συμφωνίες και συμφωνίες τελικής εμπορικής σχέσης ε, με ε, σημαντικό εμπορικό περιεχόμενο θα ακολουθήσουν και επειδή το εμπόριο είναι βασικό στοιχείο σε αυτές τις συμφωνίες ομολογώ πως προσβλέπω σε μια πιο συνεργάσιμη στάση από πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που είναι αρμόδια ευθείας για αυτές τις συμφωνίες ιστορικής σχέσης και συνεργασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Εμίλιο Μενέντες. Παρακαλώ Εμίλιο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορώ όπως και εσείς να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά σας και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να επεκταθώ περαιτέρω διότι δηλώσατε ρητά το πρόβλημα. Συμφωνώ απόλυτα για αυτό το οποίο κάναμε προηγούμενα, δηλαδή να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία. Επιτρέψτε μου να πω εν συντομία πως ορισμένες φορές θα ήταν σκόπιμο το σώμα μας να κρατάει και ενός λεπτού σιγή για την ε, απεχθή στάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλα τραγικά γεγονότα όπως ε, αυτό της άρνησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει το δόγμα προστασίας για τα όσα συμβαίνουν στην Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι και το γεγονό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε ακόμα και μετά από τα όσα είπε ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλεία ε, του ΟΗΕ και όλα τα υπόλοιπα όργανα για να αποδεχθεί αυτό τα οποία συνέβησαν μέχρι τώρα και αυτά τα οποία συνεχίζουν να συμβαίνουν. Τα λέω αυτά για λόγους αξιοπρέπειας. Ελπίζω να το συμμερίζονται οι συνάδελφοι. Δεν έχω πολλά να πω σχετικά με αυτή την πρόταση. Ακούσαμε τι αιτιολογίες σας και θα ζητήσω από την Επιτροπή να αποτανθεί στην αρμόδια ουσία. Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου το Κοινοβούλιο να μπορέσει να εγκρίνει αυτήν την συμφωνία και να υπενθυμίσω πως υπάρχουν ε, ικανοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Είτε το δούμε από πλευράς καθαρά εμπορικής, όπως ε, εξήγησατε και εσείς, επειδή είμαστε η αρμόδια Επιτροπή, αλλά και από πλευράς διεθνών σχέσεων ε, του Κοινοβουλίου. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω αυτό λόγω των όσων συμβαίνουν στην Βόρεια Αφρική. Διότι αν μπορούμε στην ε, Βόρεια Αφρική να απαγιώσουμε όχι μόνο την ε, πολιτική κατάσταση αλλά και την πολιτική που θα προκύψει από μια Αίγυπτο η οποία θα ε, βαθίζει προς τον εκδημοκρατισμό μια Τίνιδα που θα, την Ισία συγγνώμη, που θα συνεχίσει και αυτή να εκδημοκρατίζεται το, το Ιράκ να τονίσω ότι έχει δυναμωθεί από δημοκρατικής ε, πλευράς και όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε θα πρέπει να εγκριθεί αυτή η συμφωνία, να προωθηθεί και να μπορέσουμε να δομήσουμε την πολιτική, εμπορική και οικονομική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ. Δεδομένων των ε, συνθήκων νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Επιθυμεί κάποιο συνάδελφο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συμφωνώ με το σημαντικό ζήτημα αυτής της εκθέσεως και νομίζω ότι αυτή είναι και μία από τις ευθύνες της Επιτροπής μας να καταστούμε πιο ενεργοί, πιο δραστήριοι στο ζήτημα των Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με τον Ιράκ. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω πως αυτή η συμφωνία δεν είναι μια εμπορική προτιμησιακή συμφωνία και προβλέπει κάποια περαιτέρω στοιχεία σε ό,τι αφορά τις κρατικές προμήθειες και τις επενδύσεις. Και έχω κάποιες αμφιβολίες και ε, αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο περί εμπορίου είναι στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε προκειμένου να βοηθήσουμε το Ιράκ να βρει έναν νέο τρόπο για να αναδιαρθρώσει την οικονομία του. Δεν θα πρέπει να δούμε λοιπόν μόνο το θέμα της αγωνιστικότητας από Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τι μπορούμε να προσφέρουμε στους Ιρακινούς ώστε να είναι ενεργοί εταίροι στο πλαίσιο μιας ε, διμερούς σχέσης και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, Κομισιόν να σκεφτεί περαιτέρω τι θα μπορούσε να συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια οικοδόμησης ε, εταιρική σχέσης. Ίσως θα καταθέσω μια τροπολογία προκειμένου να σας ε, βοηθήσω. Ευχαριστώ. Το και Σαΐφη το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάιφη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την παρένθεση που άνοιξε ο συνάδελφος. Προσωπικά, εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει και βρίσκω απόλυτα λυπηρό, για να μην πω αξιολύπητο, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί καταρχήν το Ιράκ έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε επιτέλους να διαδραματίσει ένα πολιτικό ρόλο μετά δε αυτά, μετά δε αυτά που έλαβαν χώρα στην Τινησία και την Αίγυπτο και θα πάει στο τέλος της εβδομάδας μια αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στην οποία θα συμμετέχω και εγώ νομίζω ότι στέλνουμε ένα πολύ κακό πολιτικό μήνυμα στην περιοχή αυτή. Μετά από τα γεγονότα αυτά τα οποία ε, λαμβάνουν χώρα μπορεί στο τέλος της εβδομάδας να είμαστε θεατές μια σφαγής στη Λιβύη. Είναι πραγματικά λυπηρό το ότι δεν έχουμε το πολιτικό θάρρος που θα έπρεπε να έχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, συμφωνώ με τους συναδέλφους, οι οποίοι έλαβαν το λόγο, είναι απόλυτα ανεπαρκής η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη Βόρεια Αφρική. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν άλλες γεωπολιτικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε που μας έχουν υποσκελήσει πλήρως. Κρίμα αυτό για τις φιλοδοξίες της συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Σάιφη στο σημείο αυτό. Τώρα για τα διαδικαστικά ζητήματα. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι ότι θα πρέπει να τη συζητήσουμε επιπλέον στη συνεδρίαση των συντονιστών. Είναι πια μια παράδοση να είναι παραπεταμένη η Επιτροπή μας από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και να παραγνωρίζεται. Και δεν λαμβάνονται υπόψη στα σοβαρά οι αρμοδιότητές μας. Γίνονται τέτοιες βίαιες παρεμβάσεις, μπαίνουν στα χωράφια μας και τα καταπατούν οι άλλες επιτροπές και εγκρίνουν εκθέσεις και θέσεις οι οποίες βρίσκονται στο δικό μας τομέα αρμοδιότητας. και αυτό φυσικά αντιβαίνει με τις κατευθύνσεις που έχει ακολουθήσει πολλές φορές η Επιτροπή μας και οι οποίες έχουν επικυρωθεί και από την Ολομέλεια. Πιστεύω λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να εγείρεται το θέμα αυτό στη συνεδρία των Πρόεδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών γιατί αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στα έγγραφα Και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, προφανώς αυτό δεν ευνοεί την εργασία μας. Σας ευχαριστώ. Um, yes, um, I fully agree with you. Πλήρως σύμφωνο μαζί σας. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία να προσπαθήσω να διαλευκάνω την νομική κατάσταση σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας για τα θέματα αυτά. Έχετε στο φάκελό σας την συμφωνία. Το σημείο 3.2 είναι σε σχέση με το εμπόριο και τις επενδύσεις. Και έχουμε 72 άρθρα από 120, από το 8 στο 80 και αυτό περιλαμβάνει, το κείμενο περιλαμβάνει ορισμένα πάγια άρθρα. Αυτό σημαίνει ότι το 70% ουσιαστικά του ουσιαστικού διατακτικού σε αυτή την έκθεση είναι καθαρά θέματα εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων. Με αυτά δικά μας θέματα. Και μας παραγνωρίζουν σε αυτή την περίπτωση στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό σήμερα στη συνεδρία των συντονιστών. Ο κ. Ζάντορφ. Και εγώ ήμουν δύο φορές στο Ιράκ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι εμπειρογνώμων για τα Ιρακινά θέματα, αλλά το Ιράκ έχει τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Αν το συγκρίνουμε με άλλες αραβικές χώρες. και είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε τη σημασία του Ιράκ. Από την εμπειρία μου γνωρίζω, παραγωγός χάρη, ότι ένα από τα σημεία δυναμίας της Ιρακινής οικονομίας είναι η υποδομή. Το συνδροδομικό δίκτυο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και έχουν καταστραφεί πολλά σημεία διασύνδεσης. Υπάρχει μια ευκαιρία λοιπόν για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές υποδομών και υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες για την μεταφορά διασωτερικών υδατίνων οδών. Έχουμε δύο μεγάλους ποταμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στην εποχή του Σαντάμ Χουσέιν διότι το προεδρικό του μέγαρο ήταν στις όχθες αυτών των δύο ποταμών. Το Ιράκ διαθέτει επίσης τεράστιους φυσικούς πόρους. Έχει ε, άμμο, κοιτάσματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την παραγωγή ιάλου και παρά τον ανταγωνισμό άλλων χωρών έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ίαλο σε πολύ καλές τιμές και να τον, να την εξάγουν σε άλλες χώρες. και είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στο Ιράκ. Υπάρχουν και άλλες ε, ε, βιομηχανικές δραστηριότητες πέραν της χρήσης της ε, άμμου ή αλλουργίας για την παραγωγή ή άλλου. Υπήρχε ένα εργοστάσιο για τρακτέρ το οποίο δεν είχε πλήρως ολοκληρωθεί και υπάρχει στη Ραμάντα ένα εργοστάσιο παραγωγής κεραμικών ειδών που μπορεί να εξάγει και στο εξωτερικό. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να τα καταγράψουμε αυτά στο ενεργητικό του βιομηχανικού δυναμικού του Ιράκ ώστε όλα <coughs> αυτά τα οποία λέγονται στο, στην προσούρα μας δεν είναι επαρκή. Μπορούμε να διερευνήσουμε και άλλες δυνατότητες. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ο Εμίλιος θέλει να πει κάτι. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι προφανώς ευχαριστώ την κυρία Σάφη και τον κύριο Καζάκ που συμμερίστηκαν την απόψή μου <clears throat> και χαίρομαι πάρα πολύ και είναι τιμή μου να ακούω τα σχόλιά τους. Και στον κύριο Σόλτς επίσης θέλω να ευχαριστήσω, ο οποίος έχει παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα αυτά. Και επίσης και ο τελευταίος ομιλητής έδειξε και αυτός τόσο ενδιαφέρον όσο και ο κύριος Σόλτς και δέχομαι με μεγάλη χαρά τις προτάσεις του. Ευχαριστώ θα ακούσουμε και κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντελαγουισίγια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που ακούσαμε για την ε, συνεργασία. Υπάρχει ένα τμήμα συνεργασίας με το Ιράκ όπου προβλέπεται η υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης διάφορους τομείς κατ' της συμφωνίας. Υπάρχει αυτή η πτυχή δηλαδή. Τώρα, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση αυτή τη ε, συμφωνία, ε, προφανώ δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει του 2011 στο μέτρο που διαπραγματευτήκαμε για τη συμφωνία το 2008 και 2009. Και ε, έπρεπε να λάβουμε υπόψη την ε, μέγιστη δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι Ιρακινοί για τη διακυβέρνηση της χώρας και χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε υπό αυτές τις συνθήκες. Προσπαθήσαμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ε, προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Η διοικητική ικανότητα των ε, Ιρακινών ήταν ελάχιστη. Δεν υπήρχαν τελωνιακοί δασμοί, δεν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα δεν είχαν κανένα μέσο στη διάθεσή τους. Οπότε κληθήκαμε να προσαρμόσουμε την συμφωνία στην κατάσταση που επικρατούσε στο Ιράκ, η οποία πόρα πήγε από τη σημερινή και άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη συμφωνία να ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι η επόμενη συνεδρίαση αυτού του μήνα μέχρι το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 12 και 13 ε, Απριλίου. Ε, τώρα ας περάσουμε στο σημείο 5, εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα. και για τη θέσπιση άδεια εξαγωγή καθώ και μέτρων εισαγωγή και διαμετακόμιση για πυροβόλα, πυροβόλα όπλα. Ο εισηγητή μα είναι ο Σαλβατόρε Γιακολίνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, σήμερα, τροπολογίες που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής μας, καθώς και τα μέλη τη Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, ε, γιατί η οποία επιτροπή εκδίδει και γνωμοδότηση για την έκθεσή μας. Σαλβατόρη Γιακολίνο. Εδώ είμαι πρόεδρε. Να, απέναντί μου. Κοίταζα σε λάθος σημείο για να σας εντοπίσω. Ευχαριστώ. Ήδη συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2010. πάνω στην η πρώτη συνάντηση στην οποία εξετάζουμε τις τροπολογίες. Το κείμενο αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Εθνών για τα πυροβόλα όπλα καθώς επίσης και τη θέσπιση άδειας εξαγωγής αλλά και εισαγωγής. Αυτό το φάκελος ε, όλο αυτό το θέμα έλαβε 67 τροπολογίες ε, και έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που περιλάμβανε 33 τροπολογίες. Πολλές από τις τροπολογίες ε, της ΛΥΜΠΕ είναι τροπολογίε τι οποίε θα έξαμε στην Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να διακρίνουμε δύο είδη τροπολογιών. Η πρώτη προσπαθεί να απλουστεύσει την διαδικασία καθιστώντας πιο ευέλικτες ε, τις διαδικασίες για τους ενδιαφερόμενους. Αυτές τις τροπολογίες τις έχουν καταθέσει ένας ικανός αριθμός ε, συναδέλφων και αφετέρου Υπάρχει μια, ένα, άλλη πτυχή η οποία συνδέεται με την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα σημείο από το οποίο η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, θα μπορούσε να παρέμβει φροντίζοντας να περιορίσω αυτή την πρώτη μου παρέμβαση σε κάποιες συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τις δύο κατηγορίες θα ήθελα να ξεκινήσω από το άρθρο 2 το οποίο αφορά στους ορισμούς και επί το οποίο έχουν γίνει κάποιες τροπολογίες εγώ είχα κάνει διάκριση τα μέρη και τα βασικά εξαρτήματα. Θεωρώ ότι αυτή η στάση οδηγούσε σε μια διευκρίνηση περαιτέρω του ζητήματος και ήταν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. για Αναφέρουμε ιδιαίτερα στην, τροπολογία, στην οδηγία 51 του 98 ε, στο άρθρο 5 σε ό,τι αφορά τις άδειες και εδώ Ενδεχομένω θα πρέπει να υπάρξει κάποια συμβαστική τροπολογία προκειμένου να περιορίσουμε τους χρόνους αναμονής προτείνοντας 60 ε, μέρες προθεσμία όπως προτείνουν και κάποιοι συνάδελφοι. Το άρθρο 7 είναι κεντρική σημασίας και αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, που μπορούν να αναλάβουν ε, κάποιοι χρήστες πυροβόλων όπλων από πλευράς κυνηγών και αθλητών. είναι άτομα τα οποία εισέρχονται, ασκούν αυτή τη δραστηριότητα και εισέρχονται στο κράτος διαμονής και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η άδεια κυνηγού ή η άδεια όπλου κατοχής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενισχύ. Και υπάρχει και η παράγραφος 4 όπου οι κυνηγοί δεν ε, δεν κυκλοφορούν μόνο σε ένα κράτος μέλος, κράτος διαμονής, αλλά ε, και διασυνοριακά κάτι το οποίο όμως δεν ε, περιέχει τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Τώρα, κάτι ακόμα, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά και στο άρθρο 19 αλλά και στο άρθρο 20. Το πρώτο αφορά τις προθεσμίες που βλέπονται για την αναθεώρηση του κειμένου. Θα προτείνει αιτία, άλλοι προτείνουν ετία. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες περί αυτού τώρα. Σε ό,τι φορά τη θέση σε ισχύ, η Κομισιόν έχει προτείνει 4 μήνες, άλλες τροπολογίες μιλάνε για 36 μήνες. Εγώ είχα επαναπροτείνει έξι μήνες. Γίνεται πεπισμένος ότι σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξευρεθεί μια ε, ισορροπημένη λύση έτσι ώστε το νομοθέτημα να μπορέσει να επιτρέψει και μια αναθεώρησή του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και θα μπορούσαμε αυτούς τους έξι μήνες να τους ε, αυξήσουμε σε ένα πιο ικανό διάστημα. Αυτές, Πρόεδρε, είναι οι παρατηρήσεις από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Αν μου δώσετε τη δυνατότητα, θα ήθελα να μπορέσω να ολοκληρώσω και να σταγάγω τα συμπεράσματα. Υπαρχόντων τροπολογιών από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η συγγήτρια της Επιτροπής αυτής ήταν η κυρία Ματιού. Δεν ξέρω αν είναι παρούσα εδώ σήμερα. Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μεταξύ μας. Ο κύριος Φιόνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με διάφορους συναδέλφους υποβάλαμε από κοινού μια σειρά τροπολογιών με στόχο να απλουστεύσουμε την νομοθεσία ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική. Θεωρούμε ότι είναι περιβολικά γραφειοκρατική διαδικασία και δεν εξυπηρετεί το αρχικό στόχο της πρότασης. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και ελπίζω η συγητής ε, κ. Γιακολίνο να με ακούσει με προσοχή και να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μου. Ε, τροπολογία 60. Ε, για ποιο πράγμα δηλαδή χρειάζεται κάποιος άδεια. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό πέρα από τα όπλα να μιλήσουμε και για τα πυρομαχικά. Ε, αν ε, θέλει πάει κάποιος ε, να κυνηγήσει, παραδείγματος χάρη σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται κάποια ειδική άδεια για τα όπλα και τα πυρομαχικά. Θεωρώ ότι είναι παράλογο να χρειάζεται ξεχωριστή άδεια για τα πυρομαχικά. Μία μία άδεια και για τα δύο. Αυτή είναι η τροπολογία 60. Μετά για το άρθρο 7 Μπορείτε κύριε Σιγητά να δείτε και την ε, τροπολογία 63 και 64. Εγώ θεωρώ ότι έχουν κέρια σημασία και πάλι ο στόχος είναι να πλουστευτεί η πρόταση μέσα στο ίδιο πνεύμα. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της κοινοποίησης, τα όσα προβλέπονται στην πρόταση, δηλαδή για την κοινοποίηση Όταν ε, ε, είναι κάποιος σε μια χώρα όπου δεν διαμένει και δεν έχει άδεια οπλοφορίας κατάλαβα καλά πρέπει να αποσταλεί κοινοποίηση αν κάποιος φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στο σημείο που ε, φεύγει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη χώρα στην οποία βρίσκεται θα πρέπει να κάνει την κοινοποίηση. Μα ποια γραφειοκρατία. Ε, καλύτερα είναι να απλουστεύσουμε περαιτέρω τη διαδικασία. Επίσης με τον κύριο Γιακολίν έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και το θέμα του ορισμού, των ορισμών. Τα είπαμε και με τον Πρόεδρο. Ε, οι τροπολογίες 77 και 78 παραδείγματος χάρη σε άλλους κανονισμούς περιγράφουμε τα πάντα ως σύνολα αλλά και τα μέρη που συναποτελούν το σύνολο. Οπότε δεν πρέπει να προσαρμόσουμε ε, τους ε, ορισμούς ή εν πάση περιπτώσει να ευθυγραμμιστούμε ε, με τους υπόλοιπους ε, κανονισμούς με αυτά που ισχύουν εκεί πέρα σχετικά με τους ορισμούς και τα εξαρτήματα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν καλά σημεία μέσα στην πρόταση, αλλά υπάρχουν και πολύ χακέ τροπολογίε, όπω η 74 για την απλουστευμένη διαδικασία για αυτού που χρειάζονται περισσότερο τι άδειε. Ε, δηλαδή αυτού που ασχολούνται με τον αθλητισμό, με ε, τους, για του κυνηγού, ε, παραδείγματο χάρη. Αυτή είναι η πρώτη που θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια τέτοια απλουστευμένη διαδικασία. Είναι εντελώς παράλογη η τροπολογία 74. Επίσης η τροπολογία 68 για την διαμετακόμιση. Εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις βάσει των οποίων θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος αυτήν την άδεια, το διαβατήριο, το ενιαίο ή την εθνική άδεια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ισχύσει παντού μια ενιαία διάταξη να έχουμε μία ε, άδεια. Φανταστείτε τώρα κάποιος από την Ελλάδα ε, φτάνει στα ε, σουηδικά τελωνία και πρέπει να εξηγήσει τι λέει μέσα η άδεια, μπορεί να λέει οτιδήποτε στα ελληνικά. Μπορεί να είναι η κάρτα τη βιβλιοθήκη για να δανείζεται βιβλία στη βιβλιοθήκη. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν είναι δυνατόν. Αν υπάρχει όμω μια ευρωπαϊκή άδεια, αρκεί. Αυτά λέμε στην τροπολογία 67. Αρκεί επίσης κάποιο ε, να δείξει ε, μία φορά την άδειά του, όχι κάθε φορά που φτάνει σε ένα αεροδρόμιο ή σε κάποιο έλεγχο. Ε, Εμεί, ε, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε, δεν έχουμε απευθεία πτήσει. Ε, περνάμε από την Κοπενχάγη, από τη Φραγκφούρτη για να ε, πάμε οπουδήποτε. Αλλά, συγγνώμη, κάθε φορά που θα διερχόμαστε από μία χώρα επειδή έχουμε μία διπλή πτήση, θα πρέπει να δείχνουμε την άδεια μία φορά. αρκεί. μπορεί να σας φαίνονται λεπτομέρειες όλα αυτά, αλλά εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Thank you. Now... Ευχαριστώ. Η Ελίζαπεθ Κόστιγκερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που λέει ο κύριος Φέλνερ και να αναφερθώ στο άρθρο 7. Έχουμε ήδη μια άδεια ευρωπαϊκή για τα πυροβόλα όπλα και όλα τα υπόλοιπα εθνικά έγγραφα για την αθλητική χρήση πυροβόλων όπλων, επομένως δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε και περισσότερη γραφειοκρατία. Όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια τρίτη χώρα με τα όπλα αυτά, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλα προβλήματα για τους αθλητές και σκοπευτές. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για το έργο του γιατί νομίζω ότι θα μπορέσουμε χάρη σε αυτήν την έκθεση να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με ενδεχόμενε μικρέ τροπολογίε και μόνο. Ευχαριστώ κύριε Σλάνγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα της γραφειοκρατίας για τους σκοπευτές και τους κυνηγούς δεν θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο αυτής της οδηγίας. Η ουσία αυτής της οδηγίας είναι ακριβώ το θέμα του πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τα πυροβόλα όπλα ή καλύτερα πώς μπορεί να εμποδίσει την λαθρεμπορία πυροβόλων όπλων. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα της οδηγίας. Για το δεύτερο αυτό θέμα της ε, απλοποίησης των διαδικασιών για τους κυνηγούς και τους ε, σκοπευτές, τους αθλητές αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σκεφτούμε πώς θα το απλοποιήσουμε, αλλά θα πρέπει να είναι μια διάταξη η οποία θα είναι στεγανή, θα είναι επαρκώς καλύπτουσα τα προβλήματα αυτά και όχι να δημιουργήσει παραθυράκια για να διευκολύνει το λαθρεμπόριο των πυροβόρων όπλων. Επομένως, είναι πάρα πολύ καλή και θετική αντιμετώπιση του εισηγητή και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί της φάσης αυτής. Thank you. Uh, σας ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ρίξω νερό στο κρασί σας και εγώ πιστεύω ότι το κέντρο αυτής της οδηγίας δεν είναι φυσικά η αθλητική χρήση των πυροβόλων όπλων αλλά η σύνολη προβληματική σε σχέση με τα πυροβόλα όπλα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να εστιάσουμε τόσο στο πρόβλημα και στο φόβο της γραφειοκρατίας, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε στο δημόσιο χώρο τα πυροβόλα όπλα. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τα πυροβόλα όπλα. Τουλάχιστον αυτή είναι η στάση της Κομισιόν. Και δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ εκπροσωπώ απόλυτα αυτό το οποίο είναι η απόψη της ομάδας μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον κίνδυνο των ατυχημάτων, των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν στις κοινωνίες μας, οπότε δημιουργείται και μεγάλη κατακραυγή στις κοινωνίες μας όταν υπάρχουν ατυχήματα ενέργειες αμόκ που οδηγούν σε θανάτους πολλών ανθρώπων από άτομα τα οποία έχουν άδεια οπλοφορίας. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να τα θέσουμε στο κέντρο της εξέτασής μας για αυτή την οδηγία και να τα λάβουμε υπόψη. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια τροπολογία να καταθέσουμε ε, στο έργο του ΙΣΥΤΗ και υποστηρίζουμε απόλυτα την πρόταση της Κομισιόν. Ο κύριος και τα δύο τελευταία σημεία. Να σας πω <clears throat> απλώς, θέλω πως πω στον Μπέρντ ότι τα όπλα είναι για να σκοτώνουν. Είτε σκοτώνουν πουλιά, σπουργίτια, είτε αρκούδες, είτε ανθρώπους, είναι για να σκοτώνουν. Ανεξάρτητα από την νομοθεσία που θα σας πείσετε, πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι γίνονται πάντα ατυχήματα ό,τι και να κάνουμε εδώ στο ποδόσφαιρο με ένα αεροβόλο κάποιος πυροβόλησε ένα ποδοσφαιριστή τυχαία στο πόδι, χωρίς να το θέλει. Λοιπόν, τέτοια ατυχήματα γίνονται και όταν κάποιος παθαίνει αμόχ και αρχίζει να πυροβολεί ό,τι βλέπει μπροστά του, είναι αδύνατο να το εμποδίσουμε αυτό. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες ελέγχου όπλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς ε, ελαφρά όπλα, ακόμα και για σκοπούς αθλητικούς. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να έχει στην κατοχή του τέτοια όπλα. Ακόμα και οι αθλητές μας πρέπει να πηγαίνουν αλλού για να εκπαιδεύονται στα όπλα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα από, τους, από τα πιο ψηλά επίπεδα εγκλημάτων που έχουν πυροβόλα όπλα στην Αγγλία. Τα όπλα αυτά δεν έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχεδόν σίγουρο αυτό, έρχονται παράνομα από άλλα μέρη του κόσμου. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δυνατότητα να μπορέσει κανείς με την νομοθεσία να αποτρέψει την ε, τυχαία ή θεληματική φώνευση ανθρώπων από πυροβόλα όπλα. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι νόμοι μας είναι σωστοί, ότι τηρούνται και ότι μπορούν να εφαρμοστούν από την αστυνομία σε οποιοδήποτε κράτο για τον έλεγχο των όπλων. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίε. Και θέλω να εξηγήσω στον εισηγητή μα τη λέει τροπολογία 58. Ένα από τα προβλήματα για την παραγωγή όπλων, και μιλάω για αθλητικά όπλα εδώ, είναι η... καταρχήν ότι έχουμε πολλά νέα όπλα τα οποία έρχονται στην αγορά. Υπάρχουν πολύ λίγες εμποροπανηγύρεις για όπλα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να ζητήσουμε από όλους να πάρουν άδεια εξαγωγών για να βγάλουν τα όπλα τους και να τα πάνε εκεί. Θα χρειαζόταν τόσος χρόνος που δεν θα μπορούν να πάνε στις αρμόδιες αυτές εμπόροπανηγύρεις. είναι σημαντική βιομηχανία όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάω για εξαγωγές όπλων παράνομα, για πολεμικές ενέργειες ή για παράνομους σκοπούς. Απλώς και μόνο ο τομέας χρήσης αθλητικών όπλων είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανεί να παρουσιάζει σε εμπορικέ εκθέσει και πανηγύρι στα όπλα αυτά. Αυτό χρειάζεται συνήθω τουλάχιστον δύο μήνε για να πάρει κανεί μια άδεια για τα θέματα αυτά. Ο Κρίστοφερ Φέλεν κάλυψε τα περισσότερα ζητήματα τα οποία εγώ ήθελα να θίξω. Υπάρχει ένα ακόμα σημείο για την τροπολογία 72. για τα βασικά στοιχεία των ε, πυροβόλων όπλων και το, μνημι... το μητρό για τέτοια άτομα τα οποία έχουν κάνει σοβαρά εγκλήματα. Θα πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίσουμε εάν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να διαπράξει ένα έγκλημα. <clears throat> Έχουμε πολύ σοβαρές διατάξεις για να αποτρέψουμε την κατοχή των όπλων αυτών από τα άτομα αυτά και νομίζω ότι όταν μιλάμε για την αστυνομία, η κεντρική αστυνομική δύναμη, οι τοπικέ αστυνομίε έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν οποιονδήποτε ο οποίο έχει ένα πιστοποιητικό όπλο κατοχή. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν, γι' αυτό ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να φέρουμε αυτή την έκθεση πιο κοντά στην πραγματικότητα γιατί όσο πιο απλή νομοθεσία τόσο καλύτερα μπορεί να εφαρμοστεί και πολλοί αστυνομικοί συμφωνούν με αυτό. Είτε έχει κανείς ένα πιστοποιητικό για οπλοφορία ή δεν το έχει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν να το ελέγξουν οι αστυνομικέ δυνάμεις. Ο Κρίστοφερ κάποιος άλλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για οπλοκατοχή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσει κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειάζονται επιθεωρήσεις από την αστυνομία. <clears throat> Ήρθαν στο σπίτι μου για να μου ανανεώσουν το πιστοποιητικό. Με ρωτήσανε και πώς είναι οι συζυγικές μου σχέσεις, αν πίνω, αν κάνω χρήση ουσιών, διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν με, δεν με ρωτήσαν οδηγώ τα, τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό το βλέπουν ούτως ή άλλως από το από την άδεια κυκλοφορίας και την άδεια οδήγησης. Αλλά υπάρχει το θέμα αυτό για τα όπλα μπορεί να λυθεί με ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και όπως λέει ο Κρίστοφερ αν έρθει ένας ε, Έλληνας στην Αγγλία εκτός αν ήταν σε ορισμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε ελληνικό εστιατόριο κανείς δεν θα καταλάβαινε τι έλεγε το πιστοποιητικό του. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για το έργο του. Έχει εργαστεί σε πολύ καλή συνεργασία μαζί μου σε πολλέ άλλε περιπτώσει και είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια συμφωνία για τα κέρια θέματα σε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι ο στόχος για οποιοδήποτε όπλο θα πρέπει να είναι η προστασία των ανθρώπων. Αν ε, κάποιοι καθυστερούν στα σύνορα επειδή, έχουν, ε, επειδή οπλοφορούν, ε, συγγνώμη, είναι το τίμα που πρέπει να καταβάλουν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, για να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι. Για το πρωτόκολλο 10 των Ηνωμένων Εθνών προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και να δούμε ποιες διατάξεις θα ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τον κύριο Στέρντι και χαίρομαι που έρχονται οι αστυνομικοί και ελέγχουν τον κάθε ένα που υποβάλλει αίτημα. Έτσι θα είμαστε ασφαλείς. Πραγματικά πρέπει να προστατευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε από τα πυροβόλα γιατί ο στόχος τους είναι να τραυματίσουν και να σκοτώσουν. Γι' αυτό κατασκευάζονται. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε το κοινό, καλό είναι. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των όπλων θα πρέπει να υποστούν κάποιες καθυστερήσεις. Σας ευχαριστούμε. Ο Πίτερ Στάσνη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, αλλά επειδή έχω προσυπογράψει κάποιες τροπολογίες, ε, ήθελα κι εγώ να πάρω το λόγο για να υποστηρίξω τον Κρίστοφερ Φιέλνερ, αλλά και τον κύριο Λάγκε, ε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, διότι η ιδιοκτήτη πρέπει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια πρόληψης ε, που γίνεται. Όταν υποβάλλει κάποιος αίτηση για την άδεια, για την οπλοκατοχή, ναι, θα πρέπει να επιδιώξουμε απλούστευση ε, της διαδικασίας ε, και να εστιάσουμε την προσοχή μας αυτούς που παρανόμως έχουν στην κατοχή τους τέτοια όπλα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και ε, είναι κατανοητή η διάσταση απόψεων που υπάρχει. Αν κάποιος έχει, είναι κάτοχος αυτής της άδεια. ή μάλλον να το πω αλλιώς, ε, ο στόχος αυτής της πρότασης είναι απλούστευση της διαδικασίας και η αφαίρεση των όπλων από αυτούς που παρανόμως τα έχουν στην κατοχή τους. Μάλιστα, λέει ε, ο Πρόεδρος, ε, ο κύριος Σόλτς και πάλι και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω με μεγάλη προσοχή την συζήτηση γιατί βρίσκω ενδιαφέρουσα. Ήδη στην περιγραφή την παρουσίαση που έκανε ο εισηγητή, ε, βλέπω ότι κάποιε χώρε ακόμη δεν έχουν υπογράψει αυτό το 10ο πρωτόκολλο των Ηνωμένων ε, Εθνών. Ε, θα επιμείνω αυτή είναι η μέγιστη προτεραιότητα για λόγους δημόσιας ασφάλειας να εφαρμοστούν οι κανονισμοί και οι διατάξεις του πρωτοκόλλου. Η τσεχική δημοκρατία, Φερρυπίν, δεν έχει υπογράψει ή δεν έχουν κυρώσει Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι υποχρέωσή μας ε, να εφαρμοστεί πρώτα απ' όλα το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών γιατί έτσι ε, θα εξετάσουμε όλες ε, τις κατευθύνσεις με ποιο τρόπο μπορούμε δηλαδή να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και να τον ενισχύσουμε. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, <clears throat> πώς λέγεστε αν μπορείτε για τα πρακτικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Φάμπιο Μαρίνη από την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων και ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζοντας ε, αυτό το σχέδιο κανονισμού έλαβε υπόψη της ε, δύο βασικά στοιχεία ισορροπία και συνεκτικότητα, συνέπεια. Ε, ισορροπία όλη φορά τις απαιτήσει της ασφάλεια και την ελευθερία του εμπορίου και ισορροπία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα όσα ε, προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες αλλά και συνέπεια. Συνέπεια με τους ε, κανόνες που θέλουμε να επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που πρέπει να αντανακλούν τους, τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών. Για να το πράξουμε, κάναμε κάτι το ιδιαίτερα απλό. Είπαμε ότι ένα κράτος προτού να δώσει την άδεια για μία εξαγωγή, χρειάζεται να γνωρίζει πως η χώρα εισαγωγής με τη σειρά της έχει αδειοδοτήσει την συγκεκριμένη εισαγωγή. Και με βάση λοιπόν αυτό, αυτά τα στοιχεία θα προτείνουμε κάποιες διαδικασίες αρκετά ευέλικτες και απλές και που θα μπορέσουν να δώσουν κάποιους κοινούς κανόνες. Δηλαδή ε, το θέμα των προθεσμιών εντός των οποίων οι διοικήσεις θα πρέπει να εκδώσουν άδεια και αυτό προς ε, όφελος των πολιτών ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν κοινοί κανόνες και να αποφεύγουμε κάποιες διοικήσει να ξεπεράσουν εύλογα χρονικά διαστήματα και άλλε να εργάζονται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό θα μπορούσε να αποβεί ει βάρο ε, των επιχειρηματιών. Και υπάρχει και το ζήτημα της ε, απλοποίησης. Αυτό ε, που και ορισμένοι βουλευτές, ότι δηλαδή χρειάζεται να πλήξουμε τον παράνομο εμπόριο και όχι όσους νομίμως κατέχουν και εισάγουν όπλα. Ε, εκεί που προβλέπουμε για τους κυνηγούς, παραδείγματος χάρη και για τους αθλητές ένα ε, σύστημα με κάποιες διευκολύνσεις που ήδη προβλέπεται από την οδηγία, δηλαδή χρησιμοποίηση του διαβατηρίου του όπλου έτσι οι κυνηγοί των κρατών και οι αθλητές μπορούν να μεταβούν από μία χώρα στην άλλη μέσω της ε, υποβολής αυτού του εντύπου, μέσω της επιδείξης αυτού του εντύπου. Και αυτό ισχύει ακόμα και για τους ε, αθλητές ή κυνηγούς που θέλουν να πάνε σε τρίτη χώρα. Χρησιμοποιούν το ίδιο έγγραφο και μοναδική διαφορά και αυτό ε, συμβαίνει προς όφελος ε, του πολίτη ότι δηλαδή εάν ο κυνηγό εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση από την χώρα διαμονής τότε δεν είναι καν απαραίτητο να ζητήσει ένα διαβατήριο αρκεί να έχει την εθνική άδεια ε, κατοχής και να μπορεί να εξέλθει από τα σύνορα προς μια άλλη χώρα έτσι για να μην ε, αυξάνουμε την γραφειοκρατία και να ζητούμε συνεχώς έντυπα τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνη. Α, ε, κάτι, ο κύριος Στέρ θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Να πω ότι το πρόβλημα είναι τα παράνομα όπλα, αλλά δεν ε, είπατε πώς θα σταματήσει θα σταματήσετε την ε, κυκλοφορία των παρανόμων όπλων τα οποία φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, πολύ σωστά είπατε, θέλετε, με την πρόταση να μπορέσετε να εγγυηθείτε πως η χώρα εισαγωγής θα ε, χορηγεί την άδειά της. Κάπου άκουσα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν ε, χορηγούν άδειε ε, και αυτό που θα θέλαμε, το τελευταίο που θα θέλαμε να κάνουμε εδώ είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν ε, μπορείτε να πάτε σε κάποια έκθεση στις ΗΠΑ και άρα δεν μπορείτε να ταξιδέψετε και με το όπλο σας για να μεταβείτε στη χώρα αυτή. Χρειάζεται λοιπόν αυτή άδεια εισαγωγής, import license, δεν ξέρω πώς ε, το αναφέρει αυτό η, το έντυπο, η, το έγγραφο της νομοθεσίας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιο σχόλιο περί αυτού. Μία σύντομη απάντηση παρακαλώ από την Κομισιόν. Ναι. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αδειών εισαγωγής, περίπτωση των ΗΠΑ δεν είναι απόλυτα σωστή, διότι οι ΗΠΑ ζητούν δύο είδη άδειων για εισαγωγή. Δύο σε περίπτωση στρατιωτικού όπλου και μία σε περίπτωση μη στρατιωτικού οπλισμού. Και τα ορισμένα κράτη που έχουν τα ευρωπαϊκά στάνταρ έχουν και αυτή την ε, ίδια νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εισαχθεί ένα εμπορευματοκιβώτιο με όπλα δίχως ε, να έχει χορηγηθεί άδεια. Αλλά το πρωτόκολλο λέει τα εξή. Μας επιβάλλει τα εξή. Προκειμένου μια κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή των συμβαλωμένων μερών όπως λέει το πρωτόκολλο. Προτού να χορηγηθεί λοιπόν αυτή η άδεια μια εισαγωγή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι από την άλλη πλευρά χορηγήθηκε η άδεια εισαγωγής. Δηλαδή σε μια άδεια εξαγωγής πρέπει να αντιστοιχεί μια άδεια εισαγωγής. Ε, τώρα, αυτό που με ρωτήσατε πώς μπορείτε να πλήξετε το παράνομο εμπόριο. Μα ακριβώς το πρωτόκολλο μας το λέει. Μέσω του κριτηρίου της ανιχνευσιμότητας. Και το κριτήριο αυτό είναι αναγνωρισμένο με αυτήν την ανταλλαγή αδειών. Δηλαδή εγώ δίνω μια άδεια για εξαγωγή τη στιγμή που η άλλη πλευρά εκδίδει άδεια για εισαγωγή. Υπάρχουν μετά και άλλα ζητήματα όπως αυτό της ε, σήμανσης ε, κλπ. που αφορούν την οδηγία για την διακίνηση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποία εμείς συμπεριλαμβάνουμε τώρα για τις εξαγωγές εισηγητής. Κάποιες τελικές παρατηρήσεις παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τα σχόλια των συναδέλφων που έλαβαν το λόγο και που αναφίβολα συνέβαλαν σημαντικά και σίγουρα θα ληφθούν υπόψη σε μια περαιτέρω φάση κατά τη σύνταξη των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Τώρα πρόκειται για ένα ζήτημα αυτό της εισαγωγής και εξαγωγής όπλων ε, που αφορά ε, ποσά της τάξης του ενός δις ευρώ. <clears throat> Όπως υπενθυμήθηκε, όπως αναφέρθηκε μάλλον νωρίτερα, ορισμένα κράτη δεν έχουν ακόμα υπογράψει και κυρώσει αυτή την, αυτό το πρωτόκολλο. <clears throat> Ως εκ τούτου αυτός ο κανονισμός θέλει να καταστήσει ενία την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων προστατεύοντας ε, τους πολίτες, την ασφάλεια των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των ε, κυνηγών, των αθλητών αλλά και τα κάποια προφίλ ασφάλειας ε, και προστασίας Τώρα σε σχέση με τις επιμέρους τροπολογίες που ε, κρατήσαν οι συνάδελφοι, ανέφερα κάποια σημαντικά στοιχεία, ορισμένα αφορούν τα όπλα και τα πυρομαχικά, την ε, κοινοποίηση, τα βασικά εξαρτήματα, τα μέρη. Δεν συμφωνούμε με την τροπολογία 74, είμαστε κατά αυτής. Χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με την όρο άδεια. Η γραφειοκρατία δεν είναι ένα όριο, αλλά πρέπει να είναι μια πηγή που θα μας βοηθήσει στην εφαρμογή του κανονισμού και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κείμενο ως έχει θα συμπεριλάβει πολλά από τα σχόλια. Το πρωτόκολλο του 2001 δεν μπορούμε να περιμένουμε 3,5 χρόνια για να τεθεί σε ισχύ, όπως ε, θεωρώ ότι και θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, κάποιες επαληθεύσεις ε, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση εξισορροπημένη. Τις προσεχείς ημέρες ε, θα φροντίσουμε να συμπληρώσουμε αυτό το νομοθετικό αυτό το νομοθέτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λέει και ο κύριος Μορέιρα. 12-13 ε, Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ας Πάμε στο σημείο 6. Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανδόρας επέκταση της συμφωνίας υπομορφή ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανδόρας για τα τελωνιακά μέτρα ασφαλείας. Είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό εγώ ο ίδιος. Η απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί και το νομικό υπόβαθρο για τη σύναψη αυτού του πρωτοκόλου. Και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αναφέρω σε εσά σε ό,τι αφορά τη νομική βάση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου και εδώ έχει εκφράσει τις ανησυχίες του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναφορά στο άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο απετέλεσε αντικείμενο με, με ενός υπομνήματος στις 11 Μαρτίου από τη νομική μας υπηρεσία. Η Κομισιόν έχει προτείνει μια λύση δεν μας φαίνεται όμως ικανοποιητική και επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει, η Επιτροπή μας θα πρέπει να ζητήσει την διαβούλευση με την ε, νομική επιτροπή εφόσον το Συμβούλιο δεν θέλει να αναθεωρήσει το σχέδιο απόφασή του. Για να μην έχουμε αναπηθήματα, αποτελέσματα και δημιουργία προηγουμένων, η γραμματεία μας και εγώ ο ίδιος εξετάζουμε προσεκτικά το θέμα αυτό και εφόσον η νομική υπηρεσία είναι εδώ, θα ήθελα να τη ρωτήσω εάν θέλει να κάνει σχόλια σε σχέση με το θέμα αυτό. Πρώτου προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο ότι εμείς έχουμε θίξει το θέμα αυτό. Όχι γιατί είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το, ζήτημα, με το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά ποδή μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για το μέλλον. Θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Στην πρότασή του για μια απόφαση του Συμβουλίου, η Κομισιόν πρότεινε σε νομική βάση το άρθρο 207, το οποίο είναι η ουσιαστική νομική βάση για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι πρόβλημα, και το άρθρο 218-6α που είναι η νομική βάση για τη συνέντευξη του Κοινοβουλίου, ούτε και αυτό είναι προβληματικό, αλλά προσθέτουν και το άρθρο 218-7 της συνθήκης. Το άρθρο αυτό δημιουργεί νομικά προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χρήση του άρθρου 218.7 προϋποθέτει μία σειρά από συνθήκες. Εάν δηλαδή προτείνει η ίδια συμφωνία να υπάρχουν τροποποίησεις που γίνονται με απλοποιημένη διαδικασία με κάποιο φορέα που δημιουργεί συμφωνία. Το πρωτόκολλο αυτό το οποίο προτείνεται όμως, όπως το βλέπουμε εμείς, δεν προβλέπει καμία από αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε από τροποποίηση που γίνονται με απλοποιημένη διαδικασία, ούτε με κάποιο φορέα ο οποίος δημιουργείται από τη συμφωνία. Κατά την άποψή μας λοιπόν, η χρήση του άρθρου 218 παράγραφος 7 δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στη νομική βάση. Σε επίπεδο τώρα διαδικαστικό, γιατί η διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχετε δίκιο <clears throat> ότι η Επιτροπή Ίντα δεν μπορεί να αφαιρέσει το άρθρο αυτό ω νομική βάση, απλώ θα πρέπει να παραπέψει το θέμα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η εντύπωσή μα όμω είναι ότι πρόκειται απλώ για ένα σφάλμα, επομένω θα είχε νόημα να θίξουμε το θέμα αυτό και με το Συμβούλιο και μπορεί το Συμβούλιο να θέλει να στείλει στο Κοινοβούλιο μια διορθωτική επιστολή επί της όπου διορθώνει την νομική βάση αφαιρώντας το άρθρο 218 παράγραφος 7. Αν δεν μπορεί το Συμβούλιο να στείλει ένα τέτοιο γράμμα, για να αφαιρέσουμε το άρθρο 218 παράγραφος 7 θα πρέπει να παραπέψουμε το θέμα στην Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί έχουμε θίξει τώρα αυτό το ζήτημα, το έχουμε θίξει και μας το υπέδειξε η Γραμματεία καταρχήν. <clears throat> Αν χρησιμοποιηθεί το 218-7, τότε το Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει εξουσίες στην Κομισιόν. Αλλά μονάχα εξουσίες τροποποίησης της ε, συμφωνίας. Ενώ Εάν εμείς δεχτούμε το άρθρο 218.7, δεχόμαστε μια ευρύτερη ερμηνεία του άρθρου 218.7, όπου το Συμβούλιο εκχωρεί και άλλου είδους εξουσίες στην Κομισιόν, εδώ δεν είναι σημαντικό βέβαια, αλλά για μελλοντικέ συμφωνίε μπορεί να υπάρχει μίσον ρόλο σε αυτό το άρθρο αυτό. Παραδείγματο χάρη στη συμφωνία με την Κορέα, η εφαρμογή τη ρήτρα διαφύλαξη γίνεται με μια φυσιολογική νομοθετική διαδικασία. Αν δώσουμε όμω μια ευρία ερμηνεία του άρθρου παράγραφος 7, μπορεί το Συμβούλιο να κάνει τροποποιήσεις με εκχώρηση εξουσιών στην Κομισιόν. Γι' αυτό εμείς στήξαμε αυτό το σημείο και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Αυτό είναι το νομικό θέμα, το οποίο έχει διευκρινιστεί, αφήνοντας κατά μέρος το ερώτημα αυτό μπορούμε να αποφασίσουμε εν καιρό και για την ουσία του θέματος μπορούμε να δώσουμε την ε, σύμφωνη μας γνώμη που εξαιρεί την Ανδόρα από την υποχρέωση εφαρμογής μέτρων τελωνιακής ασφάλειας στα αγαθά τα οποία περιλαμβάνονται στο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον οι εμπλεκόμενες πλευρές μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας όπως αυτό των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν τώρα για το θέμα αυτό. Ποιος θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω. Ε, ζητείτε η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για το πρωτόκολλο αυτό. Όπως προαναφέρατε, ο στόχος ε, της πρότασης είναι το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανδόρα να συνεχιστεί ομαλά, χωρίς προσκόμματα ε, διατηρώντας όμως ε, υψηλά επίπεδα τελωνιακής ασφάλειας ε, βάσει και του πλαισίου των προτύπων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ως προς το θέμα της νομικής βάσης, ενημερώθηκε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλια που έγιναν. Παραπέμψαμε το θέμα στην νομική μας υπηρεσία και εξετάζουμε το θέμα για να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για λάθος. Η αναφορά στο άρθρο 287 λοιπόν θα δούμε αν θα παραμείνει ή αν θα διαγραφεί. Ε, σας ε, ευχαριστούμε. Η αναφορά συγγνώμη στο άρθρο 218 εδάφιο 7. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, σχόλια παρατηρήσεις. Ο Πίτερ Στάσνη από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, Είμαι αρμόδιος για αυτό το θέμα στην πολιτική μου ομάδα και θα υποστηρίξω πλήρως τον εισηγητή. The Earl of Dartmouth. Ε, ένα απλό στοιχείο θέλω να σχολιάσω. Είναι μικρή χώρα η Ανδόρα, μικρή οικονομία έχει. Παρόλα αυτά υπάρχουν τρεις μόνο χώρες που έχουν πλήρη τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μονακό, η Τουρκία και η Ανδόρα. Οπότε όταν εξετάζουμε τυχόν προηγούμενα, νομικά προηγούμενα που θα δημιουργήσουμε για την Ανδόρα, που είναι μικρή οικονομία όπως σας είπα, αλλά που είναι και προφανές, Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ε, το κατά πόσο δημιουργούμε προηγούμενο και για την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλη χώρα και μεγάλη οικονομία. Οπότε ας προσέξουμε, ε, μπορεί εκ πρώτης όψης να φαίνεται απλό το θέμα, ας προσέξουμε ποια προηγούμενα δημιουργούμε. Πρόεδρος, αντίθετα με αυτά που ισχύουν για την Τουρκία είναι και περίκλη στη χώρα η Ανδόρα και πολύ μικρή σε εμβαδόν. Ε, άλλη διαφορά με την Τουρκία. Υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, σχόλια. Όχι. Εφόσον εκρεμεί αυτό το νομικό ζήτημα που ήγηρε η νομική μας υπηρεσία, Προς το παρόν αποσύρω την ε, ημερομηνία που είχα μωρήσει για την υποβολή τροπολογιών και θα σας ενημερώσω με το που υπάρχουν εξελίξεις για αυτά τα νομικά ζητήματα. Κατόπιν, σημείο 7. Κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϊφαντουργικών ε, προϊόντων. Ο Γιάννη Ζάχραντιλ ε, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ε, είναι ο εισηγητής μας. Έχετε το σχέδιο έκθεσης στους φακέλους σας. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάργηση του κανονισμού διότι η προσκόμιση δικαιολογητικού προέλευσης θεωρείται ότι δεν έχει δεν έχει αξία. Βάσει τη συνήθου νομοθετική διαδικασία, διαβάστηκε ο φάκελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το έγγραφο εργασία από τον εισηγητή, όπου αναφέρονται και οι απόψει του. Και τώρα κατέφθασε το σχέδιο έκθεση. Γιάννη Ζαχραντήλ, που είσαι, για να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα τσεχικά. Παρακαλώ, ε, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μια προσπάθεια να είμαι σύντομος και να κάνω μια σύνοψη του προβλήματος αυτού. Έχουμε ζητήσει την κατάργηση του, κανονισμού 1541-98 και επίσης του κανονισμού, τροποποίηση του κανονισμού 3030 33/1993 93. Πρόκειται για νομικά εργαλεία τα οποία διέπουν την αναγνώριση της προέλευσης κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων στην ε, συνδυασμένη ονοματολογία τμήμα 11. Ο λόγος τώρα για τον οποίο αυτά τα εργαλεία είχαν δημιουργηθεί αφορούσε την άρση των περιορισμών για την εισαγωγή από τρίτες χώρες και ιδίως από την Κίνα. Και η η διαδικασία του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορίου είχε ήδη ε, ζητήσει την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από την ε, Κίνα. Ήδη από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 δεν ίσχυαν αυτές οι μορφές περιορισμού. Επομένως έχουμε μια πολύ καλή βάση από τα διεθνή αυτά μέσα και συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν και εγώ θα ήθελα να πω ίσως υπομορφή ηρωνίας ότι εγώ χαίρομαι να είμαι εισηγητής για ένα ζήτημα το οποίο είχε συμβάλει σε ένα πόλεμο άσκοπων κανονισμών. Νομίζω ότι με την άρση αυτών των προδιαγραφών μπορούμε επιτέλους, μπορεί επιτέλους η Κομισιόν να, να θεσπίσει μια σειρά από πιο λογικούς και επακριβείς κανόνες. Υπάρχει επίσης και η ανάγκη να υπάρξουν κανόνες για την αναγνώριση της ε, χώρας προέλευσης, για στατιστική συλλογή στοιχείων, για εκ των υστέρων έλεγχο. Δεν είναι άδεια λοιπόν τα χέρια μας, έχουμε όλη αυτή τη δυνατότητα να ασκήσουμε ελέγχους για όλα τα προϊόντα τα οποία έρχονται στην εσωτερική αγορά. Έχουμε αρκετά όπλα στην διάθεσή μας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο των εισαγωγών και για όλους αυτούς τους λόγους εγώ σας προτείνω να έχουμε μια θετική αντιμετώπιση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. From, Κάποιος από την Κομισιόν θα ήθελε να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ingrid Scharlakens από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνιακών Θεμάτων. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνατε να κάνω κάποια σχόλια εν συντομία. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη θαυμάσια αυτή η εκθεσή του όπου πράγματι κατορθώνει να θέσει στο σωστό της πλαίσιο αυτή την έκθεση. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο ουσιαστικά, ακτός από το να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία. Καταρχήν, το αντικείμενο αυτή τη πρόταση, όπω λέει και ο εισηγητή, είναι να διευκολύνει το διοικητικό, τις διοικητικές διαδικασίες και να άρει το διοικητικό άχθο των τελωνιακών διατυπώσεων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητε. Γιατί όταν ενεκρίθη ο κανονισμό αυτός υπήρχαν πράγματι υποχρεώσει. αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αιτία για, αυτός, για, αυτά για αυτούς τους κανονισμούς γιατί έχει υπάρξει ήδη η φιλελευθερωποίηση του εμπορίου υφαντουργικό. Θέλω επίση να υπογραμμίσω ότι αυτή η πρόταση δεν αλλάζει με κανένα τρόπο τι δυνατότητε που έχει ακόμα στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα σε σχέση με χώρε που δεν είναι μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και όπω τόνισε και ο εισηγητή, εξακολουθούμε να έχουμε ένα ευρύ οπλοστάσιο μέτρων ελέγχου για την διαπίστωση της προέλευσης αυτών των προϊόντων και σε περίπτωση που χωρούν <clears throat> αμφιβολίες από την πλευρά των τελωνιακών αρχών για την ορθότητα των διασαφήσεων για τα προϊόντα αυτά, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ανάγκες πρόσθετης αποδείξεως από τον εισαγωγέα. Τέλος, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή σύγχυσης, θέλω να τονίσω ότι αυτός ο κανονισμός δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στην πληροφόρηση των καταναλωτών για την οποία υπάρχουν άλλες υποεπεξεργασία νομοθετικέ προτάσει. Αυτά θέλω να πω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. <clears throat> Ναι. Η κυρία Κόπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση και της Επιτροπής και του εισηγητή στη συνέχεια για την κατάργηση ε, του κανονισμού αν δεν καταργηθεί σε αυτή τη φάση και συνεχίσει να ισχύει δημιουργεί προβλήματα συνεκτικότητας του κοινοτικού δικαίου. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον εισηγητή. Ε, στο, έργα, στο έγγραφο εργασίας που έκανε συσχετίζει τον κανονισμό αυτό με την έκθεση Μουσκαρντίνη που αφορά την ένδειξη χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες η δική μου ανάγνωση είναι ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα που δεν σχετίζονται. Πώς κατά τη γνώμη του σχετίζονται αυτοί οι δύο κανονισμοί. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το περιλάβει στο κείμενο. Κατά τα άλλα νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία και από τη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ. Uh, Κύριε Ζάχραντιλ, θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με το ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο αγαπητοί συνάδελφε. Αυτά τα δύο θέματα δεν συνάπτονται μεταξύ τους από νομική άποψη. Είναι διαφορετικές υποθέσεις. Αλλά εγώ ήθελα για λόγους πληροφόρησής σας να αναφερθώ και στα δύο και η εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε και στα δύο αυτά στοιχεία. Επομένως, η κατάργηση αυτού του νομοθετικού μέτρου με κανένα τρόπο δεν θα έχει επιπτώσει σε άλλα θέματα. Απλώς δεν υπάρχει όπως είπε η Κομισιόν κάποια επίπτωση για την πληροφόρηση των καταναλωτών. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα, απλώς είναι χρήσιμο να πληροφορούν οι συνάδελφοι για το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται αυτή η, η του κανονισμού. Any more Άλλα σχόλια. 18 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 23 ε, και 24 Μαρτίου. Ένας λιγότερο κανονισμός θα υπάρχει λοιπόν στα βιβλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείο 8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος φορέας. Ο ρόλος της πολυμερής οργανώσεις. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμεί έχουμε αποφασίσει να συμβάλλουμε με μια γνωμοδότηση και ο εισηγητής μα είναι ο Γεώργιο Λάιχφριντ. Σας δίνω, μάλλον δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα προσωπικά. Δεν μπορούσε να είναι παρόν <clears throat> στις 3 Μαρτίου, όμως μας είπε ότι θα, θα εστιάσει στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ Ό όσοι είναι γνωστό, είναι η αρμόδια επιτροπή για σχέσεις με τον ΠΟΕ. Δυστυχώς η γνωμοδότηση είναι μόνο στην Αγγλική. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε και δίνω το λόγο στον Γεώργιο Λάιχτφριντ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό είναι που ενδιαφέρεσταν είναι εδώ παρόντες όλοι και μας λέτε για την επόμενη συνεδρίαση. Αποτελεί κίνητρο, μας βοηθάτε, ξέρετε. to, Είναι μεγάλη χαρά ο συνήθως να σχολιάζει κάποιος ε, την έκθεση πρωτοβουλίας ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να ασχοληθώ με τα θέματα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου γιατί αυτό, αυτή είναι και η βασική μας αρμοδιότητα ως Επιτροπή. Το πώς εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για άλλες δραστηριότητες ένωσης ή για άλλες διεθνείς δραστηριότητες. Αν κάνετε ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες ε, του ΠΟΕ και τον ε, κανονισμό του ΟΗΕ, θα δείτε ότι θα είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Είναι ε, πάρα πολύ καλό, πάντως να εξετάσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Uh, Νομίζω ότι η συνένεση είναι ο σωστός δρόμος πρέπει να ακολουθούμε για να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ισχυρή γραμματεία στη Γενέβη. Διότι χρειάζεται ένα καλά κατερτισμένο και εξοπλισμένο προσωπικό επιτόπου για να προωθήσει τα θέματά μας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ιστορίες επιτυχίας, ας πούμε, όπως η συμμετοχή μας στον ΠΟΗ, για να εμπνευστούμε και για τη θέση της Ένωσης σε άλλους οργανισμούς. Ε, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ, ας πάρω το παράδειγμα Τη ανδόρα και της Κίνας. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό να κατέχουν ε, οι ίδια θέση σε τέτοιου διεθνεί οργανισμού όπω, ο ΠΟΕ, αλλά δεν είναι ο κατάλληλο χώρο για να το συζητήσουμε. Αφήστε που είναι και η προσωπική μου άποψη. Θα ήθελα τέλος να ε, προσέξουμε όλοι ε, τι γίνεται στις ε, διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, πώς συγχέονται τα εμπορικά με τα πολιτικά ζητήματα. Κάποια κράτη θεωρούν ότι αυτό είναι καλή ιδέα, άλλα πάλι ε, χρησιμοποιούν εμπορικής φύσεως επιχειρήματα υπάρχει διαφορά απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολύ καλά βήματα στον πω τα τελευταία χρόνια για την, ε, τον προσδιορισμό κατοφλίων, παραδείγματο χάρη. Τώρα ο Καναδάς ε, ετοιμάζεται να κάνει προσφυγή για, το, ε, για τις φώκες, για το εμπόριο προϊόντων από φώκια κατά ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου. Ε, τέτοια και άλλα παραδείγματα έχω συμπεριλάβει στην έκθεση που υποβάλλω στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Πρόεδρος, αποδείξατε ότι πάντοτε καλύτερο είναι να παρίσταται ο εισηγητής στη συζήτηση. Και σας ευχαριστούμε για τη σαφήνειά σας. Η Κομισιόν θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Η Ελιζάβεθ, η Κομισιόν, θέλει να πει κάτι. Βεβαίω, είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα σημεία που έθιξε ο εισηγητής. Τον ευχαριστούμε για τη γνωμοδότηση αυτή. Και είναι γεγονό ότι η κατάσταση στον ΠΟΕ είναι ιδανική, αλλά εδώ έχουμε μια πολύ ξεκαθαρισμένη κατάσταση για ένα οργανισμό ο οποίος αντιμετωπίζεται σε θέματα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Αυτό έχει γίνει δεκτό από όλους τους ε, εμπλεκομένους. Είναι μια πάγια κατάσταση, δεν είναι τόσο σαφής κατάσταση σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όσο στον ΠΟΕ, ιδίω σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιοτήτων. Τούτου λεχθέντος, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω του ρόλου της Κομισιόν και της Υπάτου. του εκπροσώπου και αντιπρόεδρου της Κομισιόν. Μια παρενθετική παρατήρηση η οποία υπενθυμίζει αυτά που είπε ο Ντέβιτ Μάρτιν νομίζω σήμερα το πρωί στο ατελία για το μέλλον της εμπορικής πολιτικής. Ναι, πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του ΠΟΕ για ορισμένες πτυχές, αλλά χρειάζεται να υπάρξει ο σωστός Την τρέχουσα χρονική στιγμή είναι καλύτερα να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ε, σύναψη αυτής της ε, συμφωνίας και, όχι, και μετά δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη λειτουργία του ΠΟΕ. Η Ελίζαμπεθ Κόστιγκερ από το ΕΛΚ έχει το λόγο τώρα. Μερσή κύριε Πρόεδρε, ως ε, σκιώδης εισηγήτρια από το ΕΛΚ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιχτφριντ για το σχέδιο γνωμοδότησής του και πιστεύω ότι τα τέσσερα σημεία του είναι μια πολύ καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να βασιστούμε. Εν συντομία, αναφέρθηκε από την Κομισιόν ήδη ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στον ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σαφής. Στην παράγραφο 3 σημείο 4 αναφέρθηκε εδώ και ο εισηγητής στο θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης και τις διαφάνειες των αποφάσεων που λαμβάνονται, ίσως εδώ πέρα θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη διατύπωση και από το ΕΛΚ είμαι έτοιμη να προχωρήσω σε συζητήσεις με τον εισηγητή. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την θετική συνεργασία που είχαμε με τους άλλους συναδέλφους και με τον εισηγητή. Ευχαριστώ ο Earl of Dartmouth χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ντάρτμουθ. Είναι καταθλιπτική αυτή η γνωμοδότηση γιατί περιλαμβάνει όλα τα κλισέ που ακούμε εδώ και δυόμιση χρόνια. Άλλοι τα ακούνε για 30 χρόνια και τα ξέρουν καλύτερα. Θέλω να κάνω την εξή παρατήρηση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε δίκιο. Ο ΠΟΕ μάλλον ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ είναι πολύ σαφής. Γιατί το εμπόριο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ήταν πάντα της Κομισιόν για πάρα πολύ καιρό. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1975 εμείς ως μείζον εμπορική χώρα δεν είχαμε καμία πραγματική εκπροσώπηση στον ΠΟΕ. Έχουμε εκεί μία άδεια καρέγλα ενώ το Χονγκ Κονγκ πρώην απικία έχει πλήρη εκπροσώπηση. Ως εκ τούτου υπάρχει έλλειψη παραλληλισμού μεταξύ του Ηνωμένου, των Ηνωμένων Εθνών και του ΠΟΕ. Τι νόημα έχει αυτή η αναφορά σε μία αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ΟΗΕ στη Γενέβη. Εγώ νόμιζα ότι ο ΙΕ ήταν στις Ηνωμένε Πολιτείε και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Γιατί χώρες αυτές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία που έχουν μόνιμες έδρε στο Συμβούλιο ασφαλεία. όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπροσώπησής τους μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο μικρότερη επιρροή έχουμε στο, στα Ηνωμένα Έθνη και στον όλο κόσμο. Και αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι αυτό μας δίνει μεγαλύτερη επιρροή σε παγκόσμιο <clears throat> επίπεδο. Μα αν έχετε μια μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβαθμίζει την επιρροή σας τότε έχετε λιγότερη επιρροή. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν χρειάζεται να κάνεις early για να το καταλάβει. Στο σημείο 3 αναφέρεστε στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ για να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Μα μερικές φορές οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι καλύτερο να γίνονται και κλεισμένων των θυρών και νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε και εμείς. Γιατί όταν έρχεται η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να μας συζητήσει μαζί μας γίνονται και κλεισμένων των θυρών συνήθω συζητήσεις αυτές. θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερες διαλευκάνσεις για το τι σημαίνει αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, μάλλον δεν σημαίνει τίποτα, τι θα ήθελε να σημαίνει στην πράξη αυτή η φράση. Εν τέλει, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση των μη εμπορικών θεμάτων στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ. Οι μη εμπορικέ υποθέσει. Μα το εμπόριο είναι εμπόριο. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έχει να κάνει με το εμπόριο. Για να υπάρχουν συζητήσεις για περισσότερο εμπόριο και καλύτερο εμπόριο στον ΠΟΕ δεν θα πρέπει να τις ποδηγετούμε με την πολιτική ατζέντα ορισμένων άλλων ατόμων. Ο κύριος Λάγκντορφ, λέει ο ομιλητής, μας έδωσε ένα πολύ καλό. Ο κύριος Λάιχτφριντ, η Λίχτφριντ σύμφωνα με τον ομιλητή, έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Είμαστε εδώ παρόντες σε συζητήσεις όπου έχει λεχθεί με μεγάλη σοβαρότητα από τον εκπρόσωπο του Δευτέρου Μεγάλου Πολιτικού Κόμματος στο Κοινοβούλιο ότι όλα τα συμπαρομαρτούντα της εταιρικής ε, ευθύνης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις εμπορίου. Ο κύριος Λάιχτφριντ είναι Αυστριακός και η Αυστρία έχει ανεργία 5%. Πολύ μικρό ποσοστό. Ίσως στην Αυστρία μπορείτε να δεχτείτε όλα αυτά τα προσκόμματα που έχουν να κάνουν με μη εμπορικού χαρακτήρα θέματα. Αλλά ο γείτον του κυρίου Λέιχτριτ είναι Ισπανός και στην Ισπανία η ανεργία των νέων 18-24 χρονών είναι 43%. Οι άνεργοι λοιπόν στην Ισπανία δεν μπορούν πράγματι δεν μπορούν να σκεφτούν να έχουν τέτοιου είδου μη εμπορικές ανοησίες οι οποίες εμποδίζουν τις εμπορικές συμφωνίες που θα μπορούσαν ίσως να τους δώσουν κάποια θέση εργασίας. Θέλω λοιπόν να κάνω αυτές τις παρατηρήσεις που πιστεύω ότι βρίσκονται στο κέντρο των συζητήσεων που έχουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επανέλθουμε ο εισηγητής θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τα θέματα αυτά και ίσως μπορούμε να έχουμε μία πιο ενδελεχή ανάλυση από ό,τι παρουσιάζεται στο τρέχον έγγραφο αυτό. Σας ευχαριστώ, Λεοπρόδος. Δίνω το λόγο και πάλι στον εισηγητή μας, τον κύριο Λάιχτφριντ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές οι οποίοι είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ίσως θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία από αυτά που ανέφεραν οι δύο μιλητές. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι εγώ είμαι Αυστριακός, αλλά το γεγονός ότι είμαι και Ευρωπαίος Σοσιαλδημοκράτης. Και δεν εκπροσωπώ μονάχα ε, αυστριακά συμφέροντα αλλά και θέματα τα οποία θα μπορούσαν να βρουν σύμφωνους και πολλούς ε, Βρετανούς. <clears throat> όλα αυτά τα θέματα βέβαια μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για αυτά, αλλά όλα αυτά θα αποφασιστούν με μια δημοκρατική ψηφοφορία στο τέλος. Εγώ πάντως πιστεύω ότι μια ε, άρση απαγορεύσεων για εισαγωγές δεν αφορά μονάχα τη μείωση της ε, ανεργίας στην Ισπανία έχει να κάνει και με θέματα ηθικής, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση εισαγωγών προϊόντων από φώκες. Είναι ηθικά θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε και για αυτά. Και εσείς φυσικά ακολουθείτε αυτή την άποψη γιατί υποστηρίζετε πράγματα τα οποία θεωρείτε εσείς ότι είναι από ηθική άποψη σωστά και πρέπει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται λοιπόν για τέτοια θέματα τα οποία είναι τα λεγόμενα μη εμπορικά θέματα δεν είναι μόναχα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανεργία σε κάποια χώρα. Πρόκειται για ευρύτερα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά επίσης την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου ξεκινάμε από την, το σημείο κίνησης ότι είναι μια υπόθεση μονάχα διακρατική. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Θα μπορούσε να υπάρξει μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ μια διακρατική δομή και μια διακοινοβουλευτική δομή των ΠΟΕ. Ξέρω ότι αυτό είναι μακριά από εμά. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο να οικοδομηθεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά άδικο η Ανδόρα ή το Λιχτενστάιν να έχουν το ίδιο, ίδιο ειδικό βάρος με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα. Επομένως αυτό το σημείο θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Και δεν φταίω εγώ που η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είναι στην Γενέβη και όχι στην Νέα Υόρκη. Και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θέματα τα οποία έχουν αποφασιστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι για τις συμβολές σας και ίσως <clears throat> μπορούμε να βρούμε από κοινού λύσεις σε ορισμένα από τα θέματα αυτά. Και για αυτά που είπε η κυρία Κιώστιγκερ, για τα σημεία 3 και 4, εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και αν όχι χαίρομαι για τη δυνατότητα να συζητήσω αυτά τα θέματα μαζί σας ούτως ή άλλως. <coughs> Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Φυσικά δεν το θέτω ως διαδικαστικό αλλά ως ε, ενημερωτικό προς τον ε, Βρετανό συνάδελφο. Εάν κατάλαβα καλά μιλούσατε για την ανεργία στην Ισπανία του 24% είπατε. 24 ή 42. Είπα ότι η ανεργία των νέων μεταξύ 18 και 24 είναι της τάξης του 43% περίπου. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Εν το το θέλω να προσθέσω στα όσα είπε ο συνάδελφος είναι πως η ανεργία στην Ισπανία κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλους και για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά δεν ε, εξαρτάται μόνο από αυτά που αναφέρθηκαν εδώ. Εντάξει, φυσικά η γνώμη σας ε, είναι θεμητή, αλλά εξαρτάται η ενεργεία από πάρα πολλούς παράγοντες. Και συμφωνώ με τις θέσεις το, σχετικά που αναφέρετε σχετικά με το πώς αισθάνομαστε. Εγώ αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης Ισπανικής ηθαγένειας, Ισπανικής καταγωγής. Τώρα, προθεσμία καταδεστροπολογιών 22 Μαρτίου στις 18.00. Και τώρα ας περάσουμε στο σημείο στο σημείο έλεγα 12 διότι το 11 είπαμε δεν το εξετάσουμε πρόκειται για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά εξέταση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος α είμαι εγώ εισηγητής σας και έχετε στο φάκελό σας το σχέδιο ψηφίσματος λαμβάνεις υπόψη την προγραμματισμένη επίσκεψη στον Καναδά, έχουμε καταρτήσει ένα ε, σχέδιο πρώτα ψηφίσματο και την καταθέσαμε στην Επιτροπή μας στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Επίσης, ε, προήθεται ότι θα καταθέσουμε και μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο, αλλά είναι η Κομισιόν αυτή που διαπραγματεύεται αυτές τις εμπορικές συμφωνίες και ως εκ τούτου προτείνω μια ερώτηση προς την Κομισιόν επαρκή και να αφήσουμε κατά μέρος το Συμβούλιο σε αυτή τη φάση. Σας έχει σταλεί λοιπόν το κείμενο, υπάρχει δυστυχώς μόνο στην Αγγλική. Τώρα οι διαπραγματεύσεις ε, συνεχίζονται για ε, μια συμφωνία εμπορικών σχέσεων με τον Καναδά, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. και στηρίζονται τόσο στις διαπραγματεύσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα με τον Καναδά. Σημαντική πρόοδος επαναλαμβάνω έχει επιτευχθεί και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην ε, σύναψη συμφωνίας ε, ενδεχόμενα μέχρι το τέλος ενός τότους έτους. Ε, το κείμενο περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά ζητήματα όπως πρόσβαση σε υπηρεσίες και στις δημόσιες προμήθειες και σε ε, επίπεδο επαρχιών του Καναδά, προστασία των IPR κλπ. όπως επίσης και το κεφάλαιο για την ε, αηφόρα ανάπτυξη, το ζητήματα των επενδύσεων κλπ. Ως συγητής ε, θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις σας και ως εκ τούτου έχετε το λόγο όποιος επιθυμεί να μιλήσει. Παρακαλώ τις βούλετε αγορέψει. Αυτό σημαίνει πως είστε απόλυτα σύμφωνοι με το έγγραφό μου. Ο Πίτερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες, παρακολουθούσαμε τις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε πως η ολοκλήρωση της σύναψης ε, της συμφωνίας ε, κατά του έτους ε, θα είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Υπάρχουν ε, κάποιες ανησυχίες ε, τις οποίες όλοι συμμεριζόμαστε, αλλά προσβλέπουμε σε κάποιες προτάσεις των συναδέλφων προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο αλλά και καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να μην χειροτερέψει, να μην επιδεινωθεί τουλάχιστον το κείμενο το οποίο κρίνουμε ότι θα αποτελέσει μια ικανοποιητική βάση και θα συμβάλλει θετικά στις συνολικές διαπραγματεύσεις που όπως προείπα ελπίζω να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Ο Ρόμπερ έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε τι οποίε εμεί θα θέλαμε να καταθέσουμε και θα θέλαμε να ξέρουμε πότε είναι η καταληκτική προθεσμία. Πότε πρέπει να περατωθεί η έκθεση αυτή. 21η Μαρτίου το μεσημέρι. Κύριε Λάιχτφριντ, επειδή μίλησα για τις ε, για τις φώκες προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικά ήπια η διατύπωση σε ό,τι αφορά τις φώκες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να συγκρουστούμε για τα θέματα αυτά σε επίπεδο ΠΟΕ. Ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τα θέματα αυτά προηγουμένως. Μα ο καλύτερος τρόπος να το πετύχετε αυτό είναι τροπολογίες και όχι φώκες, λέει ο πρόεδρος. Άλλα σχόλια. Ας περιμένουμε λοιπόν για τις τροπολογίες. Και πάλι καταληκτική το προθεσμία. Ξέχασα. Α, δεν ακούσαμε την Κομισιόν. Δεν δώσαμε το λόγο στην Κομισιόν. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θέλετε να πείτε τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να κάνω μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με το θέμα αυτό. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το θέμα του ΠΟΕ και των πολυμερών οργανισμών. Μιλάμε για τις φιλικές σχέσεις με τον Καναδά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού όλοι εμπόδισαν την είσοδο του Καναδά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό δεν αποτελεί βάση, κατά την άποψή μου, για φιλικές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δρούμε με τέτοιο τρόπο. Η Μεγάλη Βρετανία έχει πολύ καλές σχέσεις μέσω της κοινοπολιτείας με τον Καναδά. Τις ίδιες βασίλισσες έχουμε εξάλλου. Υπάρχει στενότατος δεσμός μεταξύ μας. Ήταν λοιπόν πολύ εχθρική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπλοκάρει την εισδοχή του Καναδά στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Και αυτό δεν θα μας βοηθήσει για να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν λανθασμένο βήμα. Μα οι Καναδοί φαίνεται δεν το θεώρησαν ότι αυτό ήταν εμπόδιο για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις του. Κατανοώ πάντως αυτό που λέτε. Ερχόμαστε λοιπόν στο κλείσιμο του ανοιχτού τμήματος και στο άνοιγμα του κλειστού τμήματος της συνεδρίασής μας. Το επόμενο τμήμα θα γίνει και κλεισμένο το θηρό Γιατί είναι συνεδρία των συντονιστών. Και ζητώ λοιπόν από όλου που δεν θα συμμετάσχουν στις συνεδρίες των συντονιστών να αποχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό.